για την εργασία που έγινε. Η μετάφραση θα είναι ε, σε λίγες εβδομάδες έτοιμη. Ζητώ συγγνώμη που δεν προλάβαμε μέχρι τώρα. Η συζήτηση για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ολοκληρώθηκε και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την συνθήκη του ΟΗΕ όσον αφορά το εμπόριο όπλων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η διεθνή Συνθήκη για τα όπλα έχει σαν στόχο να ρυθμίσει τις εκκρεμότητες σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ εύκολο να παροχετεύονται οι εξοπλισμοί σε μια παράνομη αγορά σε να αναζωπηρώνουν συγκρούσεις και να χρησιμοποιούν για ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρομοκρατία. Μπορούν να έχουν ένα ολέθριο αποτέλεσμα σε περιφερειακό επίπεδο στην ειρήνη και την ασφάλεια. Θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται κατεπηγόντως διεθνής δράση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Μέσω των διαπραγματεύσεων μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης για τα όπλα, για το εμπόριο όπλων, έχουμε την ευκαιρία να θεσπίσουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για το εμπόριο όπλων. Μπορεί αυτή η συνθήκη να κάνει το εμπόριο αυτό πιο διάφανο, πιο, να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδεσία και να αποφευθεί η παράκαμψη των κανόνων για το εμπόριο όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει πάντα ένα σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνθήκη έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τη ζωή και την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντα ότι το εμπόριο αυτό γίνεται με τον πιο υπεύθυνο τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την εκστατεία. Το ψήφισμά του 2007 στην έναρξη αυτή τη διαδικασία βοήθησε να δημιουργηθεί μια πολιτική ορμή η οποία υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή για μια συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Εγώ χαιρετίζω σήμερα την έγκριση ενό νέου ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την διάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούλιο, όπου θα διαπραγματευτεί αυτή η συνθήκη. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια. Οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμφωνήσουν τον Ιούνιο για συνολικά συμπεράσματα του Συμβουλίου για το εμπόριο όπλων, έτσι θεσπίζοντα τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαπραγμάτευση. Για να υπάρξει πραγματικό αντίκτυπο για το παγκόσμιο επίπεδο εμπόριο όπλων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η συνθήκη που θα διαπραγματευτούμε στα Ηνωμένα Έθνη θα είναι στο το πιο ισχυρή και ανθεκτική. Θα πρέπει να εξασφαλίσει αυτή η συνθήκη ότι όχι μονάχα η εξαγωγή όπλων αλλά και η διέλευση, η μεταφόρτωση και η μεσητεία των όπλων θα πρέπει να την χάνουν ελέγχους. Θα πρέπει να υπάρχει κοινή ευθύνη όλων των εμπλεκομένων για το εμπόριο όπλων. Επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα συμβατικά όπλα είναι υπό έλεγχο και όχι μονάχα τα κέρια στρατιωτικά συστήματα. Οι μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων ελαφρών όπλων μπορούν να έχουν ένα πιο αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα από μικρά από, μικρές παραδόσεις μεγάλων οπλικών συστημάτων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η συνθήκη θα περιλαμβάνει σαφείς και στεναρές παραμέτρους επί τη βάση των οποίων πρέπει να κρίνουμε τις εμπορικές συναλλαγές με όπλα. θα εξασφαλιστεί ότι οι μεταφορές όπλων και η χρήση του θα γίνεται με πλήρη σεβασμό του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Η σύμφωνη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει επίση και μια, ένα αξιόπιστο μηχανισμό εφαρμογής που ζητάει από τους κρατικούς εταίρους να θεσπίσουν εθνικά συστήματα ελέγχου για να ελέγχουν τη μεταφορά όπλων και να επιβάλλουν κυρώσεις σε μεταφορές που δεν έχουν εγκριθεί προπόντω. Τέλος, η συνθήκη αυτή θα περιλαμβάνει αξιόπιστες και σαν σαφείς μηχανισμούς ε, διαφάνειας για να υπάρξει λόγοδοσία στο παγκόσμιο εμπόριο όπλων. Η ενότητα και συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ομίλου κρατών θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να μείνουμε όμω ενωμένοι γι' αυτό. Οι υπηρεσίε μου κάνουν πολλέ προσπάθειε για να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των διαπραγματευτικών μα θέσεων, ώστε να μπορούμε να τι υπερασπιστούμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Κάνουμε επίση μια προορατική ε, προσπάθεια μαζί με του κύριου εμπλεκομένου να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Έχουμε θέσει το θέμα αυτό σε όλες μας τις ε, συναντήσεις υψηλού επίπεδου με τρίτες χώρες, με την Κίνα, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Πακιστάν και Μέξικο. Επιπλέον έχουμε κάνει μια παγκόσμια εκστρατεία προ όλε τι κατευθύνσει που να περιλαμβάνει 10 περιφερειακά σεμινάρια τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλε τι χώρε μέσα στα πλαίσια των διαποφάσεων του Συμβουλίου. Το έργο μα δεν θα τελειώσει με τη διαπραγμάτευση τη συνθήκη. Για να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο στην διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, η συνδίκη αυτή πρέπει να εφαρμοστεί και προπόντως. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μα και με την παροχή βοήθεια στι χώρε αυτέ οι οποίε είναι έτοιμε να εξασφαλίσουν αποτελεσματικού ελέγχου για τη μεταφορά όπλων, αλλά χρειάζονται τη δική μα υποστήριξη για να το κάνουν αυτό. Κυρία Άστον, περνάμε τώρα στους ε, ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Και πρώτα θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Γκάλερ, εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δέχεται τις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη και συμμετέχει σε αυτές κατά το παρελθόν υποστηρίζονταν ε, τρίτες ε, χώρες ούτως ώστε αυτόνομα να τεθεί η έλεγχο στο εμπόριο των όπλων. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο, πρέπει να υπάρξει μια ευρεία συνθήκη η οποία θα επιτρέπει ρεαλιστικό καθεστώς. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ευρεία συμμετοχή όλων των κρατών και την κάλυψη ευρέως φάσματος συμβατικών όπλων θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή να μπορεί να αντιμετωπίζει το εγκληματικό εμπόριο όπλων, το ανεξέλεγκτο. Θα πρέπει επίσης να είναι δεσμευτικό νομικά, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη ε, στο διεθνές δίκαιο. Ε, βεβαίως ο ελαφρός οπλισμός που μεταφέρεται εύκολα είναι ένα πρόβλημα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο από ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής. Ε, μου αρέσει ο ρεαλισμός σας. Πολιτικός ρεαλισμός χρειάζεται και όταν αξιολογούμε αιτήματα που θέλουν απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία και σε μη κοινοβούλια. Θα πρέπει τα, οι κυβερνήσεις να ε, συντονίζονται με τα εθνικά κοινοβούλια για τα θέματα του ελέγχου. Η επαγρύπνηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντική λειτουργία αλλά συμπληρωματική. Νομίζω ότι συνολικά θα καταφέρουμε λοιπόν και στη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη να ε, δημιουργήσουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό καθεστώς για το εμπόριο των όπλων. της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Άννα παρακαλώ. Το ψήφισμα που θα αντιμετωπίσουμε αύριο έχει να κάνει με την υπευθυνότητα, με την ασφάλεια και την πολιτική σύνδεση. Όλα αυτά ενδιαφέρουν την ανθρωπότητα για να μπορέσουμε να καταστήλουμε αυτό το λαθρεμπόριο όπλων το οποίο πλήττει τι πιο τροτέ περιοχέ του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάτι μέλη θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερο υποστηρίζοντα το πρόγραμμα δράση των ΗΠΑ κατά του παρανόμου εμπορίου ελαφρών όπλων και να αγωνιστούν στρατηγικά για μια ανθεκτική συνθήκη για το εμπόριο των όπλων που να εξασφαλίζει ότι τα όπλα τα οποία νομίμως εξάγονται και εισάγονται δεν θα παροχετεύονται για να ανατρέψουν δημοκρατικές κυβερνήσεις, για να εκμεταλλευτούν πληθυσμούς και να προωθήσουν τους πολέμους. Όλες οι πληροφορίες σε σχέση με την εξαγωγή, εισαγωγή και με τα λαμπάδευση στρατιωτικών τεχνολογιών είναι απαραίτητο να είναι γνωστή ώστε να μην οι κυβερνήσεις να γίνονται συνένοχοι των εμπόρων του θανάτου που είναι λαθρεμποριόπλων. Ε, μια συμφωνία που θα είναι αποτελεσματική θα πρέπει να θέσει ερυθρέ γραμμέ και μηχανισμού ελέγχου για την εφαρμογή τη συνθήκη αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλάει με μία μονάχα φωνή όπω η κυρία Άστον και να. Και απαραίτητα να καταλήξει σε μια κοινή θέση για όλα αυτά τα θέματα και να μπορέσει αυτή η συμφωνία να συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δικαίωμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία για δύο λεπτά παρακαλώ. Προς δεν έχουμε ξεκάθαρους κανόνες σχετικά με το εμπόριο όπλων. Ας ελπίσουμε ότι τον μήνα Ιούλιο στη Νέα Υόρκη μετά τις διαπραγματεύσεις θα έχουμε τελικά ένα σχέδιο. Είναι σημαντικό σήμερα να καταλήξουμε σε μια τελική θα έλεγα και αναλυτική συμφωνία στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής ε, να ικανοποιούνται και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κίνα, η Ινδία, η ΙΠΑ και η Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα φάση ε, έχει κάποιους κοινούς κανόνες προς τρίτες χώρες. Αυτό όμως δεν αρκεί, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να θέσω κάποια ερωτήσει. Καταρχάς, ο ιδιαίτερα πλήρης και αναλυτικός χαρακτήρας της συμφωνίας είναι σημαντικός. Αυτό που επίσης όμως έχει σημασία είναι ο έλεγχος. Έχουμε ανάγκη να υπάρξει μια δεσμευτική συμφωνία και με δεσμευτικούς υποχρεωτικούς ελέγχους. Εάν δεν υπάρξει διαφάνεια και δεν υπάρξει σωστή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα παραμείνει γράμμα κενό και σε καμία περίπτωση δεν θα εκπληρώσει τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει με τον σωστό τρόπο. Τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Ίσως αυτό το οποίο θα πω να σας φανεί κάπως ιδιόρυθμο γιατί όταν υπάρχει πόλεμος ε, κάπως αγνοούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ όμως μιλάμε για μια πιθανή συμφωνία και όταν μιλάμε για συμφωνία σημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποστέλουν όπλα σε χώρες τις οποίες κινδυνεύουν ε, να υπάρξουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ίδιος ο πόλεμος είναι κάτι τέτοιο. Κλείνοντας λοιπόν κυρία Άστον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο έχετε επιδείξει σας ευχαριστώ γιατί βοηθήσατε να προχωρήσει το θέμα αυτό με αποτελεσματικό τρόπο. η κυρία Κρόμπεκ, παρακαλώ, για 1,5 λεπτό. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση στη Συρία δείχνει γιατί χρειάζεται συνθήκη για το εμπόριο των όπλων. Η Κίνα και η Ρωσία εξάγουν πολλά όπλα στο καθεστώς Άσαντ συμβάλλοντας στο θάνατο ε, πολλών αθώων ε, παιδιών και γυναικών. Μια παγκόσμια συνθήκη για το εμπόριο θα περιορίσει και θα δυσκολέψει χώρες όπως την Κίνα και τη Ρωσία στις εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τάσεται υπέρ της μείωσης των όπλων και παγκοσμίω ε, και των πυρηνικών και ε, η συνθήκη αυτή είναι ένα πρώτο βήμα. Εμείς ε, καταθέσαμε τροπολογίες σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε για παράδειγμα μια διάκριση, δεν είναι εύκολο πια να γίνεται διάκριση μεταξύ στρατιωτικής και μη στρατιωτικής χρήσης. Ε, σε επίπεδο επιτροπής οι συνάδελφοι του ΕΛ καταψήφισαν την τροπολογία μου που αναφερόταν στην ανάγκη να υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός κατά της διαφθοράς στη συνθήκη αυτή για το εμπόριο των όπλων. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην κοινή μας θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό και ελπίζω ότι θα ψηφίσουν υπέρ της τροπολογίας οι συνάδελφοι του ΕΛΚ αύριο. Τέλος, το θέμα της ευρύτερη πρόσβασης ε, του κοινού και την πληροφόρηση για το εμπόριο στο, των όπλων. Αυτό ε, ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν τις τροπολογίες ούτως ώστε η υλοποίηση της συνθήκης να ε, να εξασφαλίσει πρόσβαση στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ ο κύριος Φανόρντεν εξ ονόματος των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα που είναι μια πολύ σωστή αξιολόγηση ενός πολύ σημαντικού θέματος. Βέβαια, η συνθήκη για το εμπόριο όπλων είναι μια εμπορική συμφωνία και δεν είναι μια συνθήκη για, την, για τον αφοπλισμό. Ο Έχω αγωνιστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για την κατάργηση και την απαγόρευση εμπορία των ναρκών κατά προσωπικού. Αυτό αφορούσε ένα συγκεκριμένο όπλο το οποίο χρησιμοποιούταν αδιακρίτως και με ολέθρια αποτελέσματα κυρίω από ομάδε ανταρτών και τρομοκράτε. Είναι σημαντικό να επεκτείνουμε αυτή τη συνθήκη και σε άλλους τομείς, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς για τον περιορισμένο στόχο αυτής της συνθήκης για το εμπόριο όπλων που δεν πρόκειται να εμποδίσει τα δικαιώματα ενός κράτου να αποφασίσει για τους δικούς του ελέγχους εξαγωγής όπλων πάντα μέσα στα πλαίσια των διεθνά, διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Είναι ο πρώτος εξαγωγέας όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν και μία από τις χώρες που προσυπέγραψαν το ψήφισμα του ΟΗΕ της 6 Δεκεμβρίου 2006 που ζήτησαν μια διεθνώς αναγνωρισμένη συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Το ψήφισμα αυτό δεν έχει μειώσει το σημαντικό ρόλο που έχουν οι αμυντικές βιομηχανίες για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία μας. Όταν συζητάμε τα θέματα αυτά, μπαίνουμε σε ευαίσθητα και σημαντικά θέματα εθνικής κυριαρχίας. Είναι κρίμα λοιπόν που το ψήφισμα αυτό ίσως αδύρυτα κινείται προς την κατεύθυνση μιας ευρωπαϊκής φεδεραλιστικής δημιουργίας αρμοδιοτήτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια συνεκτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κέρια για να μπορέσει να εγκριθεί αυτή η συνθήκη και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο ή γιατί υπάρχει κάποιος λόγος να συμμετέχει μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωριστά από τα κράτη-μέλη στη διαπραγματεύση. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να καταβάλουμε στι διπλωματικέ προσπάθειε να εξασφαλίσουμε ότι χώρε όπω η Κίνα, το Πακιστάν και η Ρωσία μπορέσουν να, θα μπορέσουν να προσυπογράψουν τα υψηλά πρότυπα που θέλουμε και όχι να σπαταλάμε τον χρόνο μα για να εναρμονίσουμε ευρωπαϊκέ θέσει που είναι πολύ πλησιωνημένε στι ΔΕ. Ας εξασφαλίσουμε να υπάρχει η προσοχή σε σχέση με τις καταχρήσεις. Το είδα αυτό στις διαπραγματεύσεις συνθήκης της ΟΤΑΒΑ. Εμείς ως, δημογρα... ως δημοκράτες αυτομαστιγωνόμαστε ενώ οι πραγματικοί καταχραστές συνεχίζουν σε να μην συμβαίνει τίποτα. Ε, Mr. John on behalf of the EFD, for one minute, please. Ο κύριος Μπάφτον εξ ονόματος του EFD για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουν υπάρξει σημαντικές αντιθέσεις στην Αμερική και στον Καναδά για την ε, συμφωνία αυτή, τη συνθήκη αυτή. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος στην εμπορία των όπλων, αλλά πρέπει να διορθωθούν οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Πάρα πολλά σπίτια στην Αμερική, πολλά νοικοκυριά έχουν όπλα και στον Καναδά επίσης, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση σε μικρά όπλα. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα όπλα λοιπόν δεν θα πιστούν από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας και σύν της άλλης υπάρχει και το θέμα της διαθεσιμότητας των όπλων στη μαύρη αγορά, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Αν υπάρξει ε, νομίζω ένα κοινό ευρωπαϊκό ε, μέτρο στον τομέα αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει θα έλεγα εισοδισμό στις αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ και των εθνικών κυβερνήσεων και θα θίξει τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτική Αριστεράς για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια το εμπόριο όπλων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την αμφίβολη ε, ε, τιμή να έχουν το 1 τρίτο του παγκοσμίου εμπορίου. 34%. Πολλέ φορέ πηγαίνουν αυτά τα ε, όπλα σε περιοχέ κρίση και σε περιοχέ όπου καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν συνολική απαγορεύση τη εμπορία όπλων, ιδίω σε περιοχέ σύγκρουση. Οι διαπραγματεύσει που γίνονται σε επίπεδο ΙΕ για τη συνθήκη για την εμπορία όπλων είναι ένα βήμα προ την σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι αυτή η η συνθήκη δεν θα καταλήξει σε ένα απέραντο χαρτοβασίλειο από πολλέ άλλε προσπάθειε στο παρελθόν. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει μια αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή, η οποία θα παραμείνει στην πολιτική ατζέντα. Το... Η συνεργασία όλων των κομμάτων στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καλό δείγμα επιτυχία και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Λυπάμαι όμω που δεν μπορέσαμε να, να αποφύγουμε μια θετική μνήα και ένα ένο προς την αμυντική βιομηχανία στην παράγραφο 2. Πιστεύουμε ότι η παρομοίωση των, ε, της αμυντικής βιομηχανίας με άλλες δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις θέσει εργασία δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Πρόκειται για μια βιομηχανία που έχει σαν μόνο στόχο το κέρδο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μετατροπή τη αμυντική βιομηχανία και χρήση των δυνατοτήτων σε άλλου τομεί. Στου ε, υπόλοιπου εγγεγραμμένου ομιλητέ και πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λίσεκ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. E, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπάτη εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να εστιάσουμε στη συνθήκη το εμπόριο όπλων τώρα με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την εστίαση στο ποδόσφαιρο. Όμως θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δραστήρια στις διμερείς ε, συνομιλίες για το εμπόριο όπλων και πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε και με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, με τη Ρωσία γιατί το εμπόριο όπλων, το ξέρουμε αυτό, πάντα ήταν αμφιλεγόμενο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευάζει, εξάγει όπλα Στη βιομηχανία αυτή δουλεύουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί μειώνονται και γι' αυτό ο κλάδος, η βιομηχανία, το κατασκευής όπλων αναζητεί νέες αγορές. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι δεν πρέπει να εξάγουμε χώρες σε περιοχές όπου υπάρχει σύγκρουση. Ούτε πρέπει τα όπλα αυτά να χρησιμοποιούνται σε αμάχους. Πρόεδρε, το νομικό κενό και η αναρχία που επικρατεί λόγω της απουσίας μιας συνθήκης εμπορίας όπλων έχει τραγικές συνέπειες, προκαλεί ανθρώπινη δυστυχία και προδίδει τις δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την προώθηση του κράτους δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης στον κόσμο. υποστηρίζουμε κατά συνέπεια στεναρά την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης νομικά δεσμευτικής και ισχυρής συνθήκης που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του εμπορίου των συμβατικών όπλων συμπεριλαμβανομένων των μικρών των κυνηγητικών και των σχετικών πυρομαχικών τους. σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διασφαλιστεί στη συνθήκη είναι η διαφάνεια της όλης διαδικασίας χωρίς διαφάνεια πράγματι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή της συνθήκης ούτε μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με την πάταξη της διαφθοράς που συχνά συνοδεύει το εμπόριο όπλων. το αρχικό κείμενο του ψηφίσματος που συζητάμε σήμερα περιείχε καλές αναφορές σε σχέση με αυτό οι οποίες όμως απαλήφθηκαν με τροπολογίες του λαϊκού κόμματος. ελπίζουμε ότι η ελομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα αναθεωρήσει αυτή τη θέση και θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξη για τη θέσπιση μια δεσμευτική συνθήκη εμπορία όπλων ένα μήνυμα που είναι κέρια σημασία εν ώψη τη κρίσιμη συνδιάσκεψη του οργανισμού ηνωμένων εθνών τον ερχόμενο μήνα. παρά τι δυσίωνε ενδείξει η συνδιάσκεψη αυτή μπορεί και πρέπει να στεφθεί με επιτυχία. σα ευχαριστώ. Ο παρακαλώ για ένα λεπτό. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να ρωτήσω τη Βαρόνια Στον. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωση σε αυτή τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια καλή συμφωνία ανάμεσα στη διακυβερνητική οργάνωση που έχει 193 μέλη κράτη και μόνο η Ζιμπάμπουε ψήφισε κατά και είναι όλοι ενωμένοι και συμφωνούν. Γιατί, ε, γιατί χρειαζόμαστε ένα υπερεθνικό εισοδιστή για να μπερδέψει τα πράγματα. Και η δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο, ε, τον οποίο μάλλον παίζει η ΙΝΤΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξοπλισμών. δεν είναι μια επιρεθνική οργάνωση και τι συνέβη από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον ε, Ιανουάριο του 2012 ε, για να επισκεφθείτε τα γραφεία της που είναι 15 λεπτά από τα δικά σας γραφεία. Τόσο μικρή σημασία έχει η ΙΝΤΑ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά τα οποία είπε η κυρία Γιάτερμάκη δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω επίσης και με τη Λέδη Άστον ότι έχουμε να κάνουμε με έναν από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι είναι, ε, θα έλεγα, ρυθμιζόμενοι σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο και έχει διασωθεί και από την οικονομική κρίση και αμφίζει. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για το 1 τρίτο του συνόλου των οπλικών εξαγωγών στον κόσμο. Στους 10 μεγαλύτερους εξαγωγείς υπάρχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες. Συνεχίζουν όμως ε, οι αλλαγές και τα προβλήματα στον χώρο αυτό λόγω των απειλών στην ειρήνη και στη δημοκρατία. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη η οποία να είναι διεθνώς δεσμευτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια συγκεκριμένη ευθύνη λοιπόν για την βελτίωση της κατάστασης. Εάν εμείς δεν μπορέσουμε να ηγηθούμε και δεν μπορέσουμε να δείξουμε αποφασιστικότητα και συντονισμό, τι μπορούμε να περιμένουμε άραγε από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να στηρίξουν πλήρως την αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών που συμμετέχει στις μελλοντικές, που θα συμμετέχει στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν άλοθη έτσι ώστε να αφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα επίπεδα των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι και οι επιφυλάξεις μας απέναντι στη Ρωσία είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη γαλλική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και όλες οι αποφάσεις για τις μεταφορές ε, όπλων και στρατιωτικών εξοπλισμών θα πρέπει να παραμείνουν ρυθμιζόμενες. Η τελευταία μου ομιλία σήμερα το απόγευμα, συγγνώμη κύρια Ήπατη εκπρόσωπος, είναι σημαντικές λεπτομέρειες αυτής της έκθεσης, αλλά σας λέω ότι είμαστε στην, στο κατόφλι μιας σημαντικής επιτυχίας για μια συνθήκη η οποία θα σταματήσει τις ανεύθυνες παραχωρήσεις και μεταφορές όπλων που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε την ευκαιρία σε μια διεθνή σύμβαση να, ε, να εμποδίσουμε μισό εκατομμύριο θανάτων το χρόνο. Πρέπει να έχουμε και μια αυτοκριτική για τις αποφάσεις μας στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων και η παροχή όπλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον άοπλων ε, διαδηλωτών στη Λιβύη, τον Μπαχρέν κτλ αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και τη σημασία του ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζήτησαν πάντα μια νομικά δεσμευτική συνθήκη. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχτήκανε τον ε, αυστηρό κώδικα της Amnesty International και θέλω να επιστήσω και την προσοχή σας στις προσπάθειες του ε, μετελθόντος ε, Ρόμπιν Κούκ, Υπουργού Εξωτερικών που ακολουθήθηκε από τον Νέτ Μίλμπαν και κατέφαλαν και οι δύο μεγάλες προσπάθειες για αυτό το ιστορικό επίθεμα. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Η κυρία Ελένα Μπασέσκου για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια και ο τομέας της άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά παίζει και ρόλο στην αναμόχλευση συγκρούσεων και αστάθειας. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ρύθμιση του εμπορίου όπλων σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει μια τροπολογία στην οποία υπογραμμίζουμε τη σημασία να υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξει σε σχέση με την αγορά όπλων. Επίση, θέλω να τονίσω τη σημασία του να υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα για να υπάρξει και η ανιχνεσιμότητα των προϊόντων από του παραγωγού μέχρι του τελικού χρήστε. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτουν μια παράγραφο του ψηφίσματος. Ένα διμερές νομικό εργαλείο θα επιτρέψει την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πιο ισχυρών αλλά και πιο διαφάνων στον τομέα αυτό και επίσης είναι αυτή η συνθήκη για να επιτύχει τους στόχους του θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες ρήτρε και πρόνοιες σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς απόδοσης ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να υπογραμμίσω και τη σημασία που επέχει το να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στην πρόληψη και την καταστολή του παράνομου εμπορίου όπλων το 2011 1.398 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε όπλα. Αυτά είναι το 2,5% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Σε μία πρόσφατη έκθεση της Oxfam καταδεικνύεται ότι τα τελευταία 12 χρόνια χώρες οι οποίες ήταν υπό εμπάρκο κατάφεραν να αγοράσουν όπλα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ευχαριστώ. Eh. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την κυρία Άστον για τα λόγια της και την κυρία Γιάχτεμάκη για την έκθεσή της. Εγώ στην θέση μου συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η Ιάννα Γκόμες και η κυρία Κοπά. Επομένως δεν θέλω να αναφερθώ επί του περιεχομένου. Απλώς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την συμφωνία αυτή και τη συνθήκη όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει σαν στόχο να θέσει κάποια τάξη σε μία μορφή εμπορίου που είναι εκτός ελέγχου. Χρειάζεται έλεγχος, υπευθυνότητα και διαφάνεια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των όπλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε εναντίον της παραγωγής όπλων. Όταν μια χώρα έχει μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά είναι πολλές φορές αντιφατικό ότι ένας υπουργό, ο οποίος ήταν υψηλός, υψηλός τέλεχος μιας ε, εταιρεία που παράγει οπλικά συστήματα να παίρνει στη συνέχεια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρέπει και εκεί να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε η παγκόσμια κοινότητα να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά και επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλάει με μία μονάχα φωνή, όχι κάθε χώρα χωριστά. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριο Πίνο Αρλάκη. Η διεθνή κοινότητα αφιερώνει πάρα πολλούς πόρους και ενέργεια σε τέτοιες ε, συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν και πάρα πολλές, επιτυχι... πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας θα έλεγα. Ταυτόχρονα τα συμβατικά όπλα και τα μικρά όπλα ε, σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες κόσμο σε αιτήσια βάση και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Αυτή η συμφωνία λοιπόν είναι μια καλή συμφωνία και οι σοσιαλδημοκράτες εκφράζουν τη λύπη τους γιατί οι χώρες μας εξακολουθούν να πολλούν πάρα πολλά όπλα σε δικτατορίες και αυταρχικά καθεστώτα. Τα ίδια κράτη-μέλη από την άλλη καθημερινά δηλώνουν την υποστήριξή τους στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά τα όπλα τα οποία πολλούν ε, θα έλεγα είναι υπεύθυνα για τις πιο προφανείς εγκληματικές ενέργειες και χρησιμοποιούνται μαζικά στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Τινησία εις βάρος των ειρηνικών διαδηλωτών. Συνεπώς λοιπόν αυτό το παράδοξο και αυτές οι αντιφάσεις θα πρέπει επιτέλους να ξεπεραστούν. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Μαυρονικόλα στην αίθουσα και θα δώσω το λόγο. Θα περάσω τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Βερονίκ Ματιό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα επικύρωσε τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με το εμπόριο των όπλων. Πρόσφατα σε έναν άλλο τομέα, αλλά εδώ είχαμε δεχθεί και την εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σχετικά με το εμπόριο όπλων. Πάντα ήμασταν κατά του παράνομου εμπορίου όπλων, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο τομέας αυτός ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνονται θα έλεγα από γραφειοκρατικές και νομικές περιοριστικές διατάξεις. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ορίσουμε σωστά τις συνθήκες ασφάλειας των πολιτών μας και το να γίνουμε πιο αυστηροί είναι κάτι το οποίο στη συγκεκριμένη φάση δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Ε, e, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στις προετοιμασίες για τη συνθήκη το κρίνω θετικά. Χρειάζεται μια ε, παγκόσμια συνθήκη σε αυτό το σημαντικό τομέα. Όμως πρέπει να τονίσω ένα πράγμα. Πολύ προσεκτικά πρέπει να σκεφτούμε τον χαρακτήρα και το εύρος της συνθήκης. Δεν πρόκειται μόνο για εξαγωγές και εισαγωγές των όπλων. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει μάλλον να δούμε τις ε, επανεξαγωγές γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ε, μέσα για να παρακάμπτονται οι διατάξεις και τα μέσα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα τεχνικά καινούργια μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ αναγνωρίζω την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει τα θέματα του εμπορίου όπλων και να επιζητήσει πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου για τη διαμετακόμιση των όπλων. Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να έχουμε ένα πιο εξελιγμένο μηχανισμό για την διανομή των όπλων και των οπλικών συστημάτων που θα να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει και έλεγχος για την περαιτέρω χρήση αυτών των όπλων και όχι μόνο να περιορίζεται στην πρώτη πώληση. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια γενική αντιμετώπιση όπου ο παραγωγός και ο διανομέας των όπλων, ιδίως για τα βαριά οπλικά συστήματα, θα έχει πλήρη έλεγχο σε σχέση με την ε, ε, συντήρηση και την παροχή ανταλλακτικών για τα όπλα αυτά. Τέτοια όπλα λοιπόν δεν θα μπορούν να μεταφέρονται σε άλλο πελάτη, μόνο να μισθώνονται. Και έτσι θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό ελέγχου όπλων και έτσι ο παραγωγός θα έχει πραγματικό έλεγχο για τη χρήση των όπλων αυτών και την χρήση τους. Ο κύριος Μέλτσερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τελευταία κατακραυγή για τα γερμανικά υποβρύχια στο, ε, στη Συρία ε, είναι αστεία, στο Ισραήλ, ε, συγγνώμη, γιατί ε, δεν πιστεύω ότι θα ήταν εξαρτημένο από εμά το Ισραήλ για να βρει ό,τι θέλει. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να ε, μην λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχει τεράστια μαύρη αγορά εδώ. Η επικείμενη διάσκεψη για την συνθήκη για τον έλεγχο μπορεί να είναι χρήσιμη για την οικοδόμηση ενός συστήματος το οποίο θα βελτιώνει τα θέματα εμπάργκο. Όμως δεν νομίζω ότι θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο όπλων. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε και όχι να κατηγορούμε τους ε, κατασκευαστές ε, όπλων και να τους επιβαρύνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καινούριε διατάξεις που δεν επιτυγχάνουν κανένας είδους αυξημένη ασφάλεια. κυρία πρέπει να αναφερθώ και σε εσά κυρία Επίτροπε. Σήμερα αυτό το θέμα που μας απασχολεί είναι η συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Θα πρέπει όμως να ατενίσουμε και τον εαυτό μας. Εμείς κάνουμε να τα ξέρουμε όλα σε σχέση με την προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε σχέση με την προστασία της νομιμότητας. Αλλά οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι αυτές οι οποίες παράγουν όπλα, δίνουν συστήματα αυτά σε τρίτες χώρες, ακόμα και χώρες όπου είναι γεγονός ότι τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν <clears throat> εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να πηγαίνουν εκεί όπλα. Και εγώ σοκάρομαι για το γεγονός ότι ένας μεγάλος παίκτη στην παγκόσμια σκηνή, η Ρωσία, δίνει όπλα στη Συρία. Και η Συρία χρησιμοποιεί αυτά τα οπλικά συστήματα για την καταστολή του πληθυσμού της και την εξολόθρευση της δημοκρατίας εκεί η εμπορία όπλων δεν θα, ήταν τόσο, δεν θα πρέπει να τόσο δύσκολο να ελεγχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά γίνονται επειδή δεν υπάρχει και σύστημα επιβολής κυρώσεων. Οι Η πάτη εκπρόσωποι της Ένωσης για τα καταληκτικά της σχόλια, κυρία Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και όλα τα μέλη για τα σχόλια που έκαναν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία για ανταλλαγές απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το σημαντικό θέμα, δηλαδή τη συνθήκη εμπορίας όπλων και πραγματικά ε, πάρα πολύ εκτιμούμε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ε, ε, προετοιμασίες στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ξέρουμε τη διαφορά μεταξύ των ε, ευθυνών και του ρόλου των κρατών μελών και των ειδικών μας και ε, σε όλα αυτά τα θέματα και στην πολιτική ασφάλεια έχουμε δεσμεύτη ότι θα ευθυγραμμιστούμε με το έργο των κρατών μελών και με αυτό που επιθυμούν τα κράτη-μέλη να κάνουμε. Επίσης ε, επιμένω ότι υπάρχει ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 27 έτσι θα αποκτήσουμε ε, κατά πολύ μεγαλύτερη δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ε, ιδιαίτερα των λεπτών θεμάτων. Ε, θα συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός δεν έχει σχέση εδώ, ευθύνεται για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Πολύ συχνά τους ε, συναντώ με πολλές ευκαιρίες. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία πρόταση ψηφίσματος και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη συρία.